Είναι ένα θέμα το οποίο επαναφέρουμε διαρκώς στο πολιτικό μας διάλογο με την Κίνα. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Έξι προτάσεις ψηφίσματος έχουμε για να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Πέρα στη συζήτηση θα ψηφίσουμε μετά από τη λήξη των συζητήσεων. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η Βερμανία και η διεξαγωγή εκλογών και η απελευθέρωση της αρχηγού της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi. Ο πρώτος συντάκτης είναι η κυρία Ντεκάιζερ για ένα μισό λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πού και πού έχουμε καλά νέα ανάμεσα στα, επίγοντα, στα κατεπήγοντα. Θα ήθελα να σας θυμίσω τη συγκίνηση που νιώσαμε όταν είδαμε να απελευθερώνεται η Aung San Suu Είναι η αλήθεια ότι έχουμε ιδιαίτερο δεσμό με αυτή την ε, αξιοσημείωτη γυναίκα που ε, πήρε το βραβείο Ζαχάροφ το 1990 και που 21 χρόνια πριν το έλαβε, στα 15 από αυτά τα έχει ζήσει φυλακισμένη. Σκεφτείτε πως μια γυναίκα πολιτικός μπορεί να ζήσει σε μια χώρα τόσο σκληρή όσο η Βυρμανία, να επιζήσει και να εξακολουθεί να αντιστέκεται. Είναι πραγματικά εξαιρετική η περίπτωση, αλλά δεν πρέπει αυτό να μας ε, κάνει να ξεχνάμε πως η απελευθέρωσή της είναι ευαίσθητη. Είναι λεπτό ζήτημα γιατί ε, ήδη είχε απελευθερωθεί και μετά τέθηκε σε κατοίκο περιορισμό. Επίσης ότι πρόκειται για ένα ομοίωμα δημοκρατίας, δεν είναι πραγματική δημοκρατία και καταπατάται η ελευθερία έκφρασης. Οι άνθρωποι όπως οι μοναχοί δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν, εμποδίστηκαν από το να ψηφίσουν. Υπάρχουν 22.000 αντιρρησίες συνείδησης φυλακισμένοι και παραμένει η χειρότερη δικτατορία του κόσμου. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από τις ε, βιρμανικές αρχές να σεβαστούν το δικαίωμα του συνεταιρίζει την ελευθερία έκφρασης, την, ελευθερία των, την απελευθέρωση μάλλον των πολιτικών κρατουμένων και εμπιστευόμαστε αυτή την ε, ε, πραγματικά εξαιρετική γυναίκα την οποία περιμένουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσει να διατηρήσει ένα πνεύμα ελευθερίας σε αυτή την τόσο ταλαιπωρημένη χώρα. Ευχαριστώ. Τρία λεπτά η κυρία Σκέικ. Ευχαριστώ. Μετά από τις ε, εκλογές η San Σανξουκή απελευθερώθηκε αφού πέρασε 25 χρόνια σε κατοίκον περιορισμό γιατί προσπεζόταν τα, τη δημοκρατία. Όπως είπε και η ίδια, η στιγμή που πάτησα το πόδι μου έξω από το σπίτι κατάλαβα ότι έφυγα από τη μία ε, φυλακή στην άλλη. Αυτή η φυλακή ονομάζεται Ιράν. Δεν θα πρέπει κανείς να ζει σε μικρές ή σε μεγάλες ε, φυλακές λόγω των ε, πεπιθήσεών του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για την υγεία και την ευημερία και την ασφάλεια της Aung San διότι κρατείται και φυλάσσεται από κρατικές υπηρεσίες. Θα πρέπει να υπάρχει ελευθερία για όλους τους πολίτες και αυτό καθορίζεται Γι' αυτό ε, το δικαίωμα το έχουν χάσει λόγω του, ε, του Θα πρέπει οποιαδήποτε κυβέρνηση να ε, έχει την νομιμότητά της βάσει της ελευθερίας των πολιτών της και κάθε πολίτης έχει δικαίωμα ε, σε κράτος δικαίου, σε σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε πραγματική διακυβέρνηση. Ο κύριος Μπίλαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όλοι εκείνοι που είχαν την ε, ψευδέστηση ότι οι λεγόμενες ε, εκλογές στην Βυρμανία ήταν γνήσιες νομίζω απεδείχθη ότι απατώντο διότι ήταν μια παροδία δημοκρατίας αυτές οι εκλογές. Μια εβδομάδα βέβαια μετά τις εκλογές απελευθερώθηκε η Ανσάν Σουτσική, αλλά παραμένουν ακόμη πάνω από 2.000 ε, κρατούμενοι στη Βυρμανία που δεν απελευθερώθηκαν. Την ίδια μέρα την οποία λάβαμε την πληροφορία από στρατιωτική ε, χούντα στη Βυρμανία για άλλη μια φορά επέβαλε περιορισμού στην ελευθερία του τύπου και έκλεισε άλλα, νέα, άλλα εννέα έντυπα. Ε, μάθαμε και την είδηση της απελευθέρωση κύρια Σανσουκή. Θα πρέπει λοιπόν να απευθύνουμε έκκληση και ιδιαίτερα προ την κυρία να πιέσει το καθεστώ τη ε, Βυρμανίας για περισσότερε ελευθερίε. Και βεβαίω ε, χαίρομαι και τιμώ την κυρία Ανσουκή για το βραβείο Ζαχάροφ. Κυρία Λόχπιλερ, παρακαλώ, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Οι εικόνες της Ανσαν Σουκί, της ηγέτητας αντιπολίτευσης στη Βυρμανία, τις στιγμές μετά την απελευθερώτησή της, είναι νομίζω χαραγμένες στη μνήμη όλων. Μια γυναίκα η οποία κρατάει ψηλά το κεφάλι μετά όλα αυτά τα χρόνια του αποκλεισμού και της απομόνωσης και που προσπαθεί να βοηθήσει τη χώρα της κάθε βήμα προς την ε, εκδημοκρατισμό και προς τη βελτίωση στην ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση των ανθρωπινών δικαιωμάτων βεβαίως είναι ευπρόσδεκτη, αλλά δεν αρκούν ακόμα. Το Σύνταγμα, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ μετά τις νέες αυτές εκλογές, επιτρέπει ε, να τίθεται υπεράνω του νόμου ο πρόεδρος του καθεστώτος, του εξασφαλίζει ατιμορρησία και του επιτρέπει κάθε είδου αυθαιρεσία. Αυτά πρέπει να τα καταδικάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω πρέπει να καταδικάσει και τι ε, απειράριθμε παραβιάσει των δικαιωμάτων, κυρίω ει βάρο των εθνοτικών μειονοτήτων, που εκδιώκονται από τη γη του, που χάνουν τη δουλειά του, που βλέπουν τα παιδιά του ε, σε ένα πεδομάζωμα να ε, συγκεντρώνονται για να εξυπηρετήσουν το στρατό τη Γερμανία. Εκείνοι οι χώρε οι οποίε έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στο καθεστώ τη Βυρμανία, όπω η Κίνα και η Ινδία, θα πρέπει να αγωνιστούν προ τον ίδιο στόχο για να υποστηριχθεί και να βελτιωθούν οι συνθήκε διαβίωση του λαού τη Βυρμανία. Και θα πρέπει οι υποσχέσει που έχουν δώσει τη διεθνή κοινότητα για την περιοχή αυτή τη Ασία να τη στηρίσουν. Όταν υπάρχουν συστηματικέ παραβιάσεις των δικαιωμάτων, πρέπει πλέον να αναλαμβάνουμε δράση. Ευχαριστώ. ένα μισή λεπτό. Σας ευχαριστώ εκλογέ. Όπω το ξέρουμε και όπω ήδη υπόθηκε εδώ στην αίθουσα, αυτέ οι εκλογέ έγιναν σε ένα κλίμα φόβου και εκφοβισμού, μια πραγματική παροδία που κατά κάποιο τρόπο εξοραίζει την εικόνα και δίνει μια πολιτική υποτίθεται ε, διάσταση στις εκλογές αυτές. Εκατομμύρια Βερμανοί αντιμετωπίζουν ε, κινδύνους, Υπάρχουν, ε, υπάρχει και αυξημένος κίνδυνος ένοπλης σύγκρουσης. Η φήμη της και απελευθέρωση της Σαν, Σαν Σουκί μας γεμίζει χαρά και ελπίδα να την δούμε και να την υποδεχτούμε εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά δεν θα πρέπει να αποσπάει την προσοχή μας από αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό στη Βυρμανία που είναι η ελευθερία ενός ολόκληρου λαού. 22.000 ε, πολιτικοί κρατούμενοι και όπως σας είπα, κλίμα εκφοβισμού και φόβο επικρατεί εκεί. Θα πρέπει λοιπόν με μέγα θάρρος να ενεργήσουμε και να μην σταυρώσουμε τα χέρια. Θα πρέπει, αξίζει την κόπο να πει κανεις οτι ότι κάποια κράτη-μέλη πρέπει να είναι πιο σταθερά στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιο συνεπή. Γιατί οι εμπορικές συναλλαγές που έχουν και εξακολουθούν να έχουν με τη Βυρμανία κάποια κράτη-μέλη η Total, ας πούμε, η πετρελαϊκή εταιρεία που αποτελεί το 7% ε, ε, των οικονομικών εσόδων της Βυρμανίας, θα πρέπει να πάψει να λειτουργεί εκεί. Ελπίζω λοιπόν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη θα επιμείνουν περισσότερο. Σας ευχαριστώ κύριο Πόσελτ για ένα λεπτό. Μιλώντα και εκ μέρου τη ε, συναδέλφου Αντρικέινε, θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου για την ε, απελευθέρωση τη θυμηθήση με το βραβείο Ζαχάροφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Σανσουκή. Αλλά υπάρχουν πολλέ χιλιάδε ακόμη κρατούμενοι στι φυλακέ ε, τη Βυρμανική Χούντα και η ίδια η χώρα, όπω υπόθηκε και νωρίτερα, ο λαό ολόκληρη τη χώρα ζει μέσα σε μια μεγάλη υπαίθρια φυλακή. Ήταν λοιπόν μόνο αισθητικού, εξοραϊστικού χαρακτήρα η επίδειξη αυτή δυνάμεως ε, του καθεστώτος ή ουσιαστικά αποδεικνύεται πως ε, οι εκλογές έφεραν το απαιτούμενο αποτέλεσμα. Θα πρέπει να πιέσουμε έτσι ώστε πράγματι να μπορέσει να έρθει εδώ το Δεκέμβριο η ε, βραβευτήσα με το, με το βραβείο Ζαχάροφ και να τιμηθεί από το Κοινοβούλιο και μετά να μπορέσει σώα και ασφαλή να επιστρέψει στην πατρίδα τη. Μόνο τότε θα πιστούμε ότι πράγματι έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα για ένα λαό που εδώ και δεκαετίε υποφέρει από μια διεφθαρμένη στρατιωτική χούντα. Ευχαριστώ και τώρα η μελετή ονόματο των πολιτικών ομάδων, ο κύριο Πρέντε για το ΕΛΚ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να χαιρετήσω την απελευθέρωση της Άγξαν Σουκί, την ε, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, ε, μετά από τόσα χρόνια κατοίκων περιορισμού. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω και την ελπίδα μου ότι αυτή η απελευθέρωση θα συνοδευτεί και από την απελευθέρωση των άνω των 2.000 πολιτικών κρατουμένων στη χώρα. Γιατί αλλιώς, ε, όπως καταλαβαίνετε, ένα προπέτασμο καπνού, είναι και τίποτα άλλο αυτή η απελευθέρωση. Επίση, θα θέλαμε να υποστηρίξουμε την Άνξανσουκι στην ε, ε, επανασύνταξη του κόμματός τη, το οποίο διαλύθηκε χωρίς λόγο το Μάιο φέτος. Πρόκειται βέβαια για ένα δύσκολο καθήκον και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι διεθνεί ε, πιέσεις, διότι η στρατιωτική χούντα δεν διερμέστηκε για κάποια δημοκρατική διαδικασία. Το αντίθετο μάλλον, οι πρόσφατες εκλογές ε, δεν ήταν ούτε ελεύθερες ούτε δίκαιες. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να ευστούμε την προσοχή μας στο θέμα αυτό. Εξ ονόματος των σοσιαλιστών για ένα λεπτό ο κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που υπάρχει ομοφωνία στο θέμα της Βερμανίας. Διάβασα τη δήλωση του Συμβουλίου, τη ε, ε, δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη δήλωση του Προέδρου μας. Όλοι χαιρέτησαν την απελευθέρωση της Άγκσαν ε, Σουκή από, από τον κατοίκον περιορισμό, αλλά όλοι καταδικάζουν το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άλλες ελευθερίες, ε, ακόμα και για την ίδια την Άγκσαν Οι εκλογές αυτές θα μπορούσαν να είναι ένα νέο ξεκίνημα για τη Βυρμανία εάν καταφέρουμε να πείσουμε την ε, στρατιωτική χούντα να απελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς κρατοποιημένους, αν τους πείσουμε να δώσουν πλήρη ελευθερία στην Αγκ Σουκή και ε, το δικαίωμα να κάνει πολιτικές δημόσιες δηλώσεις και επίσης αν η νέα κυβέρνηση αρχίσει να βελτιώνει τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων στη χώρα και επίσης να βελτιώσει τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Ίσως σε κάποια χρόνια, αν γίνουν όλα τα αυτά, θα μπορούν ίσως τα δικά μας θεσμικά όργανα να ξεκινήσουν συζητήσεις με το καθεστώς της Βερμανίας και να υπάρχει ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Όγιουλαν μάλλον δεν είναι στην αίθουσα. Ο κύριος Τσαρνέσκι, εξ ονόματος των συντηρητικών. Για ένα λεπτό. Όντως, η κυβέρνηση απελευθέρωσε μια σημαντική και γνωστή στον κόσμο προσωπικότητα για να δείξει σε όλη τη εθνική κοινότητα ότι είναι δημοκρατική και σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πίσω όμω από αυτή τη βιτρίνα, από αυτή την πρόσωψη δεν υπάρχει ουσία. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένε τροποποιήσει ή αλλαγέ στο καθεστώ. Ναι, πολύ καλό είναι που απελευθερώθηκε η κυρία Αουνσαντσουκία, αλλά πίσω από αυτό το θέατρο δεν υπάρχει άλλη ουσία παρά μόνο ότι υπάρχουν χιλιάδε ακόμη κρατουμένων σε πολύ σκληρέ συνθήκε κράτηση. Παραμένει λοιπόν επίκαιρο το θέμα των ανθρωπινών δικαιωμάτων στη Βιρμανία. Και πιστεύω πως το μήνυμα της κυρίας Αουνξαντσουκή είναι πολύ σημαντικό. Πρόκειται για ένα μήνυμα το οποίο αντιχεί σε ολόκληρη την Ασία Γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι ίδιοι αγωνιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Κίνας έχουν την Aung San Suu ως σημείο αναφοράς και είδωλο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κιουτάσου τώρα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς ζητήσαμε την απελευθέρωση της Αγκ ε, Suu επανειλημμένα από το 1990. Ε, απελευθερώθηκε τώρα η Αγκ Είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Είναι ένα θετικό βήμα. Ωστόσο δεν μπορούμε να θεωρήσουμε πως η συγκεκριμένη κατάσταση είναι λύση όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εφόσον πολλοί ακτιβιστές είναι ακόμα στην φυλακή. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχει διάταξη που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προωθήσει την ειρήνη και τη δημοκρατία δημοκρατία με κοινέ αξίε, σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατία και αξιοπρέπεια. Έχουμε καθήκον να μην περιοριστούμε στην προάσπιση αυτών των αξιών μόνο εντό τη Ένωση. Γι' αυτό έχω μια έκκληση να στείλουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύη προ του πολίτε τη ε, Βερμανία που είναι, βρίσκονται υπό την πίεση τη κυβέρνηση και καθημερινά αγωνίζονται ώστε να γίνουν σεβαστά τα βασικά του δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ταραμπέλα. Πρόεδρε, 7 Νοεμβρίου έγιναν οι πρώτες εκλογές εδώ και 20 χρόνια στη Βυρμανία. Εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε χαρή μπροστά σε μια τέτοια διαδικασία. Ωστόσο, άλλη μια φορά σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να καταδικάσουμε τη χώρα αυτή που δεν ε, κάνει τίποτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πνίγει, πνίγει και την ελευθερία έκφρασης. Ωστόσο, ε, Πώς μπορούμε να μιλάμε για επιλογή για όταν τα κόμματα αντιπολίτευσης δεν μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα, δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν ελεύθερα τον πληθυσμό. Και πάλι αναφέρομαι εδώ ότι η Βυρμανία είναι μια χώρα που δεν είναι ελεύθερη, είναι στα χέρια στρατιωτικής χούντας όπως είναι γνωστό τη Σπάση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια παγωμένη ε, δύναμη, μια εξουσία η οποία θα παραμείνει από τη στιγμή που δεν διοργανώνονται ελεύθερες ε, εκλογές. Η απελευθέρωση Σαν είναι μια χειρονομία προς τη σωστή κατεύθυνση, πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να το χαιρετήσουμε. Όμως θα χρειαστούν και άλλες ε, χειρονομίες απέναντι σε πολλού άλλους ε, πολυάριθμους ε, πολιτικούς κρατούμενου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Ελβέστρης. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή Όλοι ακόμα είμαστε υπό την επιρροή ενθουσιασμού για την απελευθέρωση της Σαν και θυμόμαστε τις εικόνες, τον κόσμο που την υποδέχθηκε, βρήκε τα παιδιά της, ε, τα έχει αφήσει μικρά και τα ξαναβρήκε ενήλικες πια. Μεγάλη χαρά για το λαό, για την αντιπολίτευση της ε, βερμανικής ε, αντιπολίτευσης. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή συνομιλητός της μας είναι η στρατιωτική χούντα που πρέπει να ξεκαθαρίσει αν αυτή η απελευθέρωση ήταν μόνο προπαγάνδα, ένα προπέντασμα καπνού ή αν είναι πράγματι ένα βήμα προς την αναγνώριση των δικαιωμάτων ελευθερίας έκφρασης και άρα και για όλους τους άλλους ε, πολιτικούς κρατούμενους στη Βερμανία ε, μια ελπίδα και ένα βήμα προς πραγματικές ελεύθερες εκλογές. Γιατί η απελευθέρωση αυτή θα πρέπει να ακολουθηθεί από ένα έντονο αίτημα προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ και τέλος ο κύριος Σόνικ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εξότιμοι κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Θυμόμαστε ακόμα νομίζω όλοι τα χρόνια εκείνα που χαιρετίζαμε και εορτάζαμε την απελευθέρωση του Λεχβαλέσα του Νέλσον Μαντέλα. Αποφυλακίσεις που έδιναν ελπίδες για ένα νέο κόσμο για έναν κόσμο στον οποίο θα υπήρχε χώρος για καταπίεση. Για έναν κόσμο που θα άλλαζαν στάση οι κυβερνήσεις. Εδώ λοιπόν με την απελευθερώση της Aung San Suu νομίζω ότι έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας γιατί κάναμε εμείς πάρα πολλές προσπάθειες, έκανε ολόκληρη η κοινότητα πολλές προσπάθειες και χωρίς αυτές τις προσπάθειες δεν είχαμε καταφέρει σήμερα να χαιρετίζουμε την απελευθέρωση της Aung San Suu Και μην ξεχνάμε ότι και στην περίπτωση των κομμουνιστικών κυβερνήσεων οι διεθνεί πιέσει ήταν αυτέ οι οποίε βοήθησαν. Γιατί ναι, είχαν συναντηθεί εκπρόσωποι των ελεύθερων κρατών με τον Λεχ Βαλένσα, είχαν πιέσει ανοιχτά τι ε, κατασταλτικές κυβερνήσει και το ίδιο θα πρέπει να γίνει και τώρα. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να έρθει η κυρία Σανξουκή στο Κοινοβούλιο. Ο κύριος Λεβαντόφσκι παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής ε, στην κυρία Άγξαν Σουκή που μόλις ε, απέκτησε την ελευθερία της κάτω από βραβείο Νόμπελ και βραβείο Ζαχάροφ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξακολουθεί να είναι ένα σύμβολο δύναμης και ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον το οποίο αξίζουν ε, οι άνθρωποι της χώρας της. Η κυρία Άγξαν Σουκή όμως θα πρέπει να έχει ελευθερία του λόγου χωρίς όρους, απεριόριστη. Και επίσης, όπως είπε και ο κύριος Πόσολ και ο κύριος Πρέσντα, υπάρχουν και ακόμα πάνω από 2.000 πολιτικοί κρατούμενοι. Θα πρέπει να απελευθερωθούν και αυτοί. Αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε μια ομελή μετάβαση προς ένα πιο δημοκρατικό σύστημα. Η Βυρμανία έκανε διεξήγαγε εκλογέ οι οποίες δεν ήταν στα πλαίσια των διεθνών προδιαγραφών, διότι δεν υπήρχε δυνατότητα να συμμετέχουν ε, κόμματα της αντιπολίτευσης. Όμως είναι αλήθεια ότι η κοινωνία της πολιτής, ε, των πολιτών κατέφερε κατά κάποιο τρόπο να οργανωθεί χωρίς βέβαια να ξεχνάμε ότι πάντα υπήρχαν προσκόμματα. Βέβαια κάποια κόμματα δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν αλλά κάποια άλλα κόμματα ακόμα και από εθνοτικές ομάδες κατάφεραν να συμμετάσχουν σε εκλογές. και η αποφασιστικότητά τους να δράξουν την ευκαιρία είναι αξιομνημόνευτη. Βέβαια, θα μπορούσε να είναι και μια ευκαιρία για μια νέα αρχή και να εισαχθεί τουλάχιστον κάποιος βαθμός πολυφωνίας ε, στο όλο σύστημα. Παρά το γεγονός ότι είναι προφανή τα ασφάλματα, εάν οι εκλογές αποτελούν την έναρξη μιας θετικής διαδικασίας, είναι κάτι ευπρόσδεκτο από πλευρά μας. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να ε, ξεκινήσει επαφές με την κυβέρνηση, ώστε οι εκλογές αυτές να αποτελέσουν μια νέα και θετική φάση για την ιστορία της χώρας. Από τούτο και στο εξή θα πρέπει να παρακολουθούμε στενά ε, τι γίνεται με το Κοινοβούλιο, κατά πόσον είναι υπόλογο προς την κοινωνία κατά πόσον ε, τα νέα όργανα θα σεβαστούν τις ανθρώπινες ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα και θα, κατά πόσον θα ξεκινήσουν νέες διαδικασίες για να σεβαστούμε τους πολίτες. Για να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην ε, χώρα θα πρέπει να υπάρχει επικοδομητικός διάλογος με όλους τους ενδιαφερομένους. Ο διάλογος αυτός θα πρέπει να θεμελιώνεται και να οδηγήσει στη μετάβαση σε ένα σύστημα δικαιοσύνης και κυβέρνησης που θα βασίζεται στο κράτος δικαίου και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να υποστηρίξει μια τέτοια διαδικασία. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας, το διάλογο και τη δέσμευσή μας, τους διάβλους των Ηνωμένων Εθνών, περιοριστικά μέτρα αλλά και συνδρομή προκειμένου να βοηθήσουμε την νέα κυβέρνηση να βελτιώσει ε, τις επιδόσεις της. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, είναι ε, εντεταγμένα στα προγράμματα βοήθειας και επίσης στην κοινωνία των πολιτών και στην κυβέρνηση. Επίσης θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να επιτύχουν τους στόχους της χιλιοτίας προάγοντας τις αξίες μας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανάπτυξη, το διάλογο που θα εξακολουθήσουν να αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής μας. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση και προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Ψηφοφορίες παρακαλώ. Πρώτα έχω